Σας ευχαριστώ. Ξέρω ότι είναι μια πάρα πολύ έντονη μέρα στο Κοινοβούλιο σήμερα με πολλές ακροάσεις. Αν θα μπορούσαν να κάτσουν παρακαλώ όλα τα μέλη. Καλημέρα σε όλους. Θέλω να καλωσορίσω την κυρία Ελσπιέτα Μπιενκόφσκα, την υποψήφια επίτροπο. Θέλω να χαιρετήσω και τον κύριο Μπούζεκ, ο οποίος είναι πρόεδρος Επιτροπής ε, Βιομηχανίας Έρευνας και Βιομηχανίας. Είναι μια κοινή συνεδρίαση, όπως ξέρετε, μεταξύ της ΙΜΚΟ και της ΙΤΡΕ και θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω τα μέλη από τις Επιτροπές ΕΜΒΙ και Γιούρι που συνδέονται με την ακρόαση αυτή και από τα μέλη της Επιτροπής Τραν Μεταφορών που έχουν προσκληθεί επίσης. Η, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς είναι αυτή που είναι αρμόδια για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, περιλαμβάνει τα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με τον εντοπισμό και την άρση ενδεχομένων φραγμών για την εφαρμογή της ενιαίας αγοράς και αυτό περιλαμβάνει και την ψηφιακή ενιαία αγορά. Η προστασία όμως των οικονομικών συμφέροντων των καταναλωτών όπως και η πολιτική και η νομοθεσία για την εφαρμογή των κανόνων της ενίας αγοράς και αυτά, αυτά περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλακείο μας. Προσβλέπουμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η προσέγγιση που θα ακολουθήσει η κυρία Μπιανκόφσκι σε αυτούς τους τομείς και πώς θα μπορέσει να βοηθήσει το έργο της δικής μας Επιτροπής και πώς η υποψήφια κύριε Επίτροπος θέλει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του τομεί αυτούς. Ελπίζουμε ότι η υποψήφια θα κατανοήσει και τις ε, ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα της Επιτροπής μας για τη μελλοντική ανάπτυξη ενιαίας αγοράς ώστε να δώσει θετικό ε, θετική βοήθεια στους καταναλωτές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης, επιχειρήσεις και στην οικονομική μεγέννηση. Και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπούζεκ για τα δικά του σχόλια. Σας ευχαριστώ κυρία Συν Πρόεδρε. Θέλω να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Θα ήθελα να δώσω ένα θερμό καλωσόρισμα στην κυρία Σβιέτα Μπιενκόφσκα, στην υποψήφιο επίτροπο. Τα μέλη του Κοινοβουλίου και από τις πέντε επιτροπές που ανέφερε η συνάδελφός μου κυρία Φόρτ πριν από δύο λεπτά, η πρόεδρος της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ, και επίσης όλοι οι εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής κοινωνίας, ε, ΜΚΟ, βιομηχανίες και φυσικά όλοι αυτοί που μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να τονίσω ότι η Επιτροπή Ήτρε είναι η Επιτροπή που είναι αρμόδια για την ε, βιομηχανία, το επιχειρήν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ένα σημαντικό τμήμα λοιπόν του χαρτοφυλακίου της κυρίας Βιενκόφσκα. Πιστεύουμε ότι θέλουμε να έχουμε μια ανταγωνιστική Ευρώπη, αλλά αυτό σημαίνει πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα, στην επικοινωνία, στα δίκτυα μεταλαμβάνευσης της γνώσης και θέματα που έχουν να κάνουν ακόμα και με την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν αυτά είναι στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Ήτρε. Αλλά μερικά από αυτά είναι τα πιο σημαντικά και αυτά βρίσκονται στο χατοφυλάκιο της κυρίας Πιενκόφσκη. Υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα πέντε χρόνια σε όλους αυτούς τους τομείς και προσδοκούμε να δούμε, να γνωρίσουμε πώς η υποψήφια κυρία Επίτροπος θέλει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Να προσθέσω κάποια τεχνικά σχόλια εξ αρχής για τη διενέργεια της ακρόασης. Η ακρόαση έχει σαν στόχο να επιτρέψει τα μέλη του Κοινοβουλίου να αποφασίσουν ποια είναι η απάντησή του σε δύο ερωτήματα. Πρώτον, αν έχει τα απαραίτητα προσόντα υποψήφιο επίτροπο για ένα μέλο του Σώματο των Επιτρόπων. Και δεύτερον, αν έχει τα απαραίτητα προσόντα για να διεκπαιρεώσει τα συγκεκριμένα καθήκοντα που τις έχουν ανατεθεί, δηλαδή το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρχαν τέσσερα διαθέσιμα έγγραφα, το βιογραφικό, η αποστολή της κυρίας Βιενκόφσκη, η δήλωση των ε, οικονομικών συμφερόντων και επίσης η, το, η επιστολή από την Επιτροπή Γιούρη και φυσικά και οι απαντήσεις στα ερωτήματα τα γραπτά των βουλευτών που έχουν μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Η διαδικασία μας είναι η συνηθισμένη, αλλά θα την επαναλάβω και πάλι. Η υποψήφια επίτροπος προσκαλείται να κάνει μια εναρκτήρια παρουσίαση που δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Θα έχει επίσης στο τέλος τη ακρόαση 5 λεπτά για μια καταληκτική παρέμβαση ή ερωτήσεις. Θα είναι 45 από τους βουλευτές, από τις διάφορες επιτροπές κυρίως όμως από την Επιτροπή ΙΜΚΟ και την Επιτροπή ΙΤΡΕ, αλλά επίσης και από τις ΕΝΒΙ, ΙΟΥΡΙ και ΤΡΑΝ. Λιγότερες ερωτήσεις για τις τελευταίες επιτροπές, γιατί είναι απλώς συνδεόμενες επιτροπές στην ακρόαση. Και θα ακολουθεί η αρχή της επιτραπέζης αντισφαίρησης, τρία λεπτά συνολικά για κάθε ερώτηση, ένα λεπτό για την ερώτηση και δύο λεπτά για την απάντηση. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τα χρονικά όρια. Πέντε λεπτά ανοχή, πέντε δευτερόλεπτα συγγνώμη, ανοχή θα έχω για το, τις ερωτήσεις των βουλευτών και λυπάμαι πάρα πολύ κυρία υποψήφια επίτροπε, αλλά εσείς θα έχετε μόνο δέκα δευτερόλεπτα ανοχή για να ξεπεράσετε το χρόνο των δύο λεπτών, γιατί θα πρέπει να κρατήσουμε το χρόνο σε κάθε ερώτηση. Έχουμε μονάχα τρεις ώρες για τις 45 ερωτήσεις. Ο πρώτος γύρος θα αφορά τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσω ότι έχουμε διερμηνία σε 23 ε, γλώσσες και επομένως ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μητρική του γλώσσα ή όποια άλλη γλώσσα επιθυμεί μεταδίδεται από την ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου στο διαδίκτυο η ακρόαση, οπότε μπορούμε πράγματι να προχωρήσουμε και να σας ζητήσω κυρία υποψήφια, υποψήφια Επίτροπε να λάβετε το λόγο για 15 λεπτά το μάξιμο.